Σας επαναλαμβάνω λοιπόν και στα αγγλικά μόνο 11 άτομα μπορείτε να ψηφίσετε. Στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποια διόρθωση, παρακαλώ απευθυνθείτε στους κλητήρες να σας δώσουν καινούριο ψηφοδέλτιο και το παλιό θα καταστραφεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Yes, okay. Uh, what Okay, okay. Uh, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, παρέμεινε η ερώτησή μου μετά από αυτές τις ε, λεπτομερείς εξηγήσεις που δώσατε. Fine, <laughs> Κυρίε ehm, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος που επιθυμεί ακόμα να ψηφίσει. Κάποιος θέλει να ψηφίσει. Ρωτάω για τρίτη φορά εάν κάποιος θέλει να ψηφίσει. Κοσοβάνιο. Ωραία. Ψήφισαν και οι ε, καταμετρητές των ψήφων. Πέρας της ψηφοφορία. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τους καταμετρητές των ψήφων να πάνε στην αίθουσα R01101 και η συνεδρίαση διακόπτεται. Θα επαναληφθεί όταν ακούσετε το κουδούνι και δείτε την ανακοίνωση στις οθόνες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως αν χρειαστεί και τρίτος γύρος ψηφοφορίας θα ξεκινήσουμε στις 7 ή 7 και μισή. Παρακαλώ μην φύγετε από το κτίριο γιατί μάλλον θα ξαναψηφίσουμε στις 7 ή στις 7.30. Οπότε μην απομακρυνθείτε από το κτίριο. Σας ευχαριστώ πολύ και διακόπτεται η συνεδρίαση.